el señor presidente. Buenos días, queridas amigas. Καλημέρα σας ε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι. Άρχεται η συνεδρίαση με το πρώτο μας σημείο σήμερα το πρωί, την έκθεση του κυρίου Deutsch για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ετήσια της έκθεση για το 2008. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον εισηγητή, τον Ταμάς Deutsch για τέσσερα λεπτά. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε της ΕΤΕΠ, κύριε Μαϊστατ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για το 2008 που είναι και το σημερινό θέμα, πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Βέβαια η έκθεση αυτή δεν περιορίζεται σε μια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το έτος 2008. Διαπιστώνουμε ότι ξεκινά μια νέα εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη θέση σε ισχύ πριν από ένα εξάμεινο της συνθήκης της Λισαβόνας και τον αντίκτυπο της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ε, που χρήζει αντιμετώπισης. Όλα αυτά στη νέα εποχή που αρχίζει με την ε, νέα συνθήκη της Λισαβόνας και το δεύτερο και τον 21ο αιώνα. Έχουμε λοιπόν ε, αυτό το ιστορικό υπόβαθρο που χρωματίζει αυτή την αιτήσια έκθεση για το 2008 και αν δούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΤΕ, διαπιστώνουμε ότι είναι πολλές. Οι δραστηριότητες της Τ.Ε.Π. Ε, για το 2008 είναι πολύ εντυπωσιακέ. Και παρά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, δεν ε, μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τη σημαντική συμβολή της ΕΤΕΠ που αντέδρασε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και άμεσα στην αντιμετώπιση της κρίσης και μάλιστα αύξησε την παροχή δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας κάθε μηχανισμό και διευκόλυνση που είχε για να προωθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να βοηθήσει τους διάφορους οικονομικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν το σχέδιο ανάκαμψης. Με τις εποπτικές ρυθμίσεις ε, δημιουργήθηκαν ε, νέες προϋποθέσεις και για την ΕΤΕΠ και νομίζω ότι ήδη από το 2008 και πριν τη θέση ισχύ της Ηθίκης Λισαβόνας έγιναν πολύ σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της εποπτείας. Στην περίοδο μετά το 2014 θα έχει να ετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ε, δράση της έναντι των μακροπεριφερειών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η ΕΤΕ μέσα από το νέο σύστημα της συνθήκης της Λισαβόνας και τη στρατηγική του 2020 θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας χάρη σε μέτρα και δανειοδοτική δραστηριότητα που θα εξυπηρετούν ακριβώς το στόχο αυτόν. Αυτό το στόχο τον έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειες. Δεν θέλω επιπλέον να υπογραμμίσω τα εξής επιμέρους ότι δηλαδή η ΕΤΕ θα πρέπει και στο μέλλον ε, ακόμη περισσότερο να δαδρά ευθυγραμμισμένα, εναρμονισμένα με τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ε, το προγράμματα όπως και οι δομές θα πρέπει να ακολουθούν ε, τους στόχους που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη έλαβε πέρυσι τη στήριξη του Κοινοβουλίου για την πολιτική αυτή. Και πιστεύουμε ότι και φέτος θα της χορηγήσει το τυποθήτο το Κοινοβούλιο, όπως άλλως το αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντόιτς. Θα δώσω τώρα το λόγο με πολύ χαρά για την παρουσία του στον κύριο Φίλιπ Μάιστατ τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε με την πρόσκληση να λάβω το λόγο εδώ στην Ολομέλεια. Κάτι που συνιστά συνέχεια μιας παράδοσης που εγκαινιάσαμε πριν από αρκετά χρόνια. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόιτς, τον εισηγητή για την πολύ ποιοτική έκθεσή του. Και εκτιμώ ιδιαίτερο που και ο κύριος Ντόιτς αλλά και άλλα μέλη της Επιτροπής, Πάρμαν, Κάλφιν, μπήκαν στον κόπο να έρθουν στη... στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να θέσουν πολύ εύστοχες και διεξοδικές ερωτήσεις. Και χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ΕΤΕΠ είναι το μόνο διεθνές χρηματοπιστωτικό όργανο που οικειοθελώς ε, είναι υπόλογο ε, και δίνει λογαριασμό σε ένα κοινοβουλευτικό όργανο και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι ουσιώδες ε, γιατί μας επιτρέπει να διενεργήσουμε την ειδική μας αποστολή και το ρόλο μας που είναι να είμαστε μεν τράπεζα, αλλά όχι μια συνηθισμένη τράπεζα, μια τράπεζα που θα εξυπηρετεί τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την ενίσχυση τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπω είπε ο κύριο Ντόιτ, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στην κρίση, να ανταπεξέλθουμε στι προκλήσει που δημιούργησε. Και από το Σεπτέμβριο του 2008, την πτώχευση τη Lehman Brothers, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, ΕΚΟΦΗΝ, μα ζήτησε να αυξήσουμε το σύνολο των δανείων μα προ την, πραγματική οικονομία. Ανασκουμποθήκαμε λοιπόν προσπαθώντα να ανταποκριθούμε σε αυτή τη σύσταση του Συμβουλίου και είμαστε σε θέση να πούμε ότι ανταπεξήλθαμε στις υποχρεώσεις μας γιατί το 2008 το, από 58 δισεκατομμύρια περάσαμε σε 79 δισεκατομμύρια δηλαδή αύξηση κατά 37% του συνόλου των δανείων που χορηγούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η εντυπωσιακή αύξηση του όγκου των δανείων μας αφορούσε κυρίως τους τρου, τρεις που και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όρισαν ως προτεραιότητες. Ο πρώτος τομέας ήταν ε, μια ιδιαίτερη προσπάθεια για τις περιοχές και τις χώρες που επλήγησαν δρυμύτατα από την κρίση και αυτή η αύξηση αφορά κυρίως τις ε, περιφέρειες και περιοχές σύγκλησης όπως λέμε και ιδιαίτερα στοχεύσαμε ορισμένες χώρες που ιδιαίτερα το 2009 αντιμετώπισαν ε, ορισμένες δυσκολίες. Για παράδειγμα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Ρουμανία. Δώσαμε δάνεια προς τις χώρες αυτές άνευ προηγουμένου. Και φέτος θα καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες για την Ελλάδα. Πήγα την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα και από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση συμφωνήσαμε ότι θα αυξήσουμε αισθητά τον όγκο των δανείων μας προς την Ελλάδα ως ένδειξη υποστήριξης ε, και συμβολή στην ε, γενική προσπάθεια που γίνεται για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας. Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας είναι η υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυξήσαμε τα δάνειά μας προς τις τράπεζες ώστε να συνεχίσουν να δανείζουν αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με, νέα, με νέα προϊόντα προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερος έλεγχος της αποτελεσματικής χρήσης των κονδύλιων αυτών. Πάνω από 12 δισεκατομμύρια δανείσαμε πέρυσι στις τράπεζες για δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ο τρίτος άξονας προτεραιότητας που μας ζητήσατε ε, να υπογραμμίσουμε είναι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Πέρυσι ε, δώσαμε περίπου 17 δισεκατομμύρια χρηματοδοτώντας ε, σχέδια και προγράμματα που συμβάλλουν ε, άμεσα στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το 2009 ανταπαξήλθαμε στην αποστολή μας και συμβάλαμε τα μάλα στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης. Φυσικά θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και θα ήθελα να αναφερθώ στις τρεις μείζονες προκλήσεις που έχουμε για το μέλλον. Η πρώτη πρόκληση είναι φυσικά και το επισήμανε πολύ σωστά ο εισηγητής είναι να υλοποιήσουμε αυτές τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ΕΤΕΠ θα συμβάλλουμε και εμείς στην ε, υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική εγκαινίασε αυτή τη νέα στρατηγική που αυτή τη στιγμή εξετάζεται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και η ΕΤΕΠ είναι έτοιμη να συμβάλλει στη υλοποίηση αυτής της στρατηγικής με καινοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που θα αυξήσουν το αποτέλεσμα αυτής της μόχλευσης ορισμένων ε, κοινοτικών κονδυλίων και ταμείων. Οπότε θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι κοινοί μηχανισμοί μεταξύ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερη σημαντική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ε, ανανέωση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση που εντάσσεται πλήρως ε, στα συμπεράσματα της Επιτροπής των Σοφών υπό την Προεδρία του κυρίου Κοντεσού. Και το κεντρικό σημείο αυτής της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Γιατί ξέρετε ότι χαίρομαι εγγύησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, ε, δραστηριότητες που εντάσσονται στην εξωτερική εντολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια πλούστευση και μια εναρμόνιση αυτής της εξωτερικής εντολής. Και μάλιστα τα 2 δισεκατομμύρια που τέθηκα στο αποθεματικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αφιερωθούν σε σχέδια που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και αυτό με φέρνει στην τρίτη πρόκληση που θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω για το μέλλον, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα να συμβάλλει προκειμένου να τηρηθούν οι υποσχέσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κοπενχάγη. Γιατί εκεί αναλάβαμε πολύ σημαντικές δεσμεύσεις ε, για να υποστηρίξουμε το Fast Track Financing και στο πλαίσιο αυτό η τράπεζά μας που έχει σημαντική εμπειρογνωμοσύνη για το θέμα αυτό μπορεί να συμβάλλει τα μάλα στην υλοποίηση αυτού του μηχανισμού. Γι' αυτό προτείναμε σε συνεργασία με άλλους εθνικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς να ιδρύσουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για καλύτερο συντονισμό και πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση των διαφόρων αναπτυξιακών σχεδίων. Και μάλιστα ήδη μια γερμανική τράπεζα έδειξε ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή και ευελπιστούμε ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλλουμε στην ε, εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Αυτές είναι οι βασικότερες μας προκλήσεις για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος Όλη Ρεν για να μας παρουσιάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόιτς για την εξαίρετη έκθεσή του. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μέιστερ και να τον καλωσορίσω και εγώ εδώ στην Ολομέλεια που και για τις προσπάθειες που έκανε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να βοηθήσει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας κάτω από τις έκτακτες συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, κάναμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ανταποκρίθηκε αμέσως και επιτάχυνε την ε, δανειοδότησή της και μπόρεσε να το κάνει αυτό ακόμα και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Αυξήθηκε ο όγκος λοιπόν των δανείων σε δύο κυρίως τομείς που πιστεύουμε εμείς ότι είναι πολύ σημαντική και ξέρω ότι συμφωνεί με αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για τις προτεραιότητές μας, κυρίως υπέρ των μικρών και μεσαίων ε, επιχειρήσεων και υπέρ τη καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Έγιναν επενδύσεις λοιπόν σε αυτούς τους τομεί, αλλά και στι περιοχές σύγκληση που επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Επιπλέον, η ΕΤΕ σε κοινή πρωτοβουλία και με την Παγκόσμια Τράπεζα και με την Τράπεζα Αναπτύξεως στήριξε τον οικονομικό τομέα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που επίσης πέρασαν δύσκολους καιρούς με την οικονομική κρίση. Η ΕΤΕ θα έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στην εφαρμογή της στρατηγικής για το 2020, στηρίζοντας επενδύσεις στις υποδομές, στις πράσινες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, θα βοηθήσει με άλλα οικονομικά μέσα και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περιοχές σύγκλησης όπου η ΕΤΕ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να ενισχυθεί η απορρόφηση των κονδυλίων από τα διαφορετικά ταμεία. Επίσης, στο εξωτερικό είμαι πολύ ευχαριστημένος για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση όσον αφορά το έργο της ΕΤΕ που κατέληξε στην εγγύηση που προσφέρει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ΕΤΕ και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Η έκθεση που εξετάζεται σήμερα περιλαμβάνει και πολύ καλές προτάσεις για την ευθυγράμμιση των εξωτερικών δράσεων της ΕΤΕ με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πώς θα ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΤΕ και την Τράπεζα Αναπτύξεως. Αυτό φαίνεται από τις εκθέσεις τις σχετικές του 2007. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε καλύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο τραπεζών. Και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι και οι δύο τράπεζες έχουν καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά την ε, συνεργασία που θα αποτελέσει και τη βάση για τριμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα, θα αντικαταστήσει τις περιφερειακές συμφωνίες. Το αποτέλεσμα πάντως είναι η νομοθετική πρόταση που μόλις υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τροποποίηση της ε, αποστολής όσον αφορά το υπόλοιπο των δημοσιονομικών προοπτικών. Πιστεύω ότι θα βρείτε την πρόταση καλά ισορροπημένη και ότι ακολουθεί τις συστάσεις και τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την εξωτερική εντολή σε στόχους ε, κλειδί, σε πολιτικές κλειδί, όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές, οι υποδομές και ο ιδιωτικός τομέας, η ανάπτυξη τοπικά του ιδιωτικού τομέα. Επίσης υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα και την ανάπτυξη Οπότε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κύριε Πρόεδρε, εν καταλήδη, Κατακλείδη θέλουμε επικοδομητική συνεργασία και συζητήσεις μαζί σας, αλλά και με το Συμβούλιο και αυτό προσδοκάμε τους επόμενου μήνες. Ελπίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα όσον αφορά την εντολή για εξωτερικές δράσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να πετύχει τους εξωτερικούς πολιτικούς της στόχους. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Επιτροπερέν, τώρα εκ μέρου τη Οικονομική Επιτροπή για δύο λεπτά η συνάδελφο Νίκη Γκέρι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. είμαι συνάδελφοι. Η Επιτροπή Οικονομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων έχει διατυπώσει τη γνωμοδότησή της με ε, τις θέσεις της, όπου επισημαίνει τα θετικά αποτελέσματα ως προς τη διαχείριση της κρίσης, τις καλές επιδόσεις της ΕΤΕΠ και την προσπάθεια ε, πάνω απ' όλα για εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας ώστε να αντιμετωπιστούν ε, οι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Δάνεια λοιπόν σε λογικά επίπεδα, με λογικά επιτόκια. Αυτό είναι ο στόχο, ώστε να μπορούν και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να ανθέξουν τη δυνατότητα αυτή. Γιατί, γιατί κάναμε αυτή την επιλογή, διότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι ο κύριος, η, η, ε, κύρια πηγή δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να εξασφαλίζουμε νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και οι τράπεζες ανα το χρήμα και αξιοποιώντας τους σε αυτούς τους στόχους μπορούν να προσφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος στις κοινωνίες μας. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε στην, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ και από την άλλη να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια αυτών των δραστηριοτήτων. Ξέρετε βεβαίως ότι ε, τα προβλήματα τα αντιμετωπίσαν κυρίως ε, οι χώρες οι οποίες μάλλον τη βοήθεια ε, την προσελκύουν κυρίω οι χώρε οι οποίε επλήγησαν περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει και τι περιφερειακέ αλλά και τι ε, τράπεζε αποταμίευση, τα ταμιευτήρια δηλαδή, να τι περιλάβουμε στην υποστήριξη που θα προσφέρουμε. Και επίσης τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως εταίροι θα πρέπει να χαρακτηρίζουν 20% των ποσών που διαθέτουν ως χρηματοδότηση απευθυνόμενη ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπα, καλά, λοιπόν, έχει, όπως είπα ήδη λοιπόν έχει ανταποκριθεί καλά η ε, ΕΤΕΠ στην κρίση, έχει προσφέρει πολύ σημαντική αρρωγή και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει με την ίδια πολιτική και στο μέλλον. Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και για ένα λεπτό. Το λόγο έχει η κυρία Κάντενμπαχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκ μέρους τη Επιτροπής θα Περιφερειακών Υποθέσεων, θα ήθελα, θα καταρχάς να ευχαριστώ ε, τη συνάδελφο για την έκθεση. Βεβαίω χαιρετίζουμε την ε, αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕΠ και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχύσει με την στάση της και τα δανειά της κοινωνική και οικονομική συνοχή και τον στόχο της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης χαιρετίζουμε τη χορήγηση 21 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά ως δάνεια, 41 δηλαδή του συνολικού ποσού που χορηγεί ε, για στο, ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απευθύνονταν ιδιαίτερα στους στόχους της σύγκλησης και τα μέτρα της ΕΤΕΠ ε, βλέπουμε με ικανοποίηση ότι ακολουθούν τους στόχους που έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τους στόχους της σύγκλησης. Ελπίζουμε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει έτσι. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στους ομιλητές εκ μέρους των κοινοβουλευτικών ομάδων. Και για δύο λεπτά πρώτος θα είναι ο Ζαμπιέρ Οντί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, Χαιρετίζω την παρουσία σας εδώ κύριε Πρόεδρε Μέστατ και ιδιαίτερο στην προσωπική μου χαρά που σας βλέπω εδώ διότι είχα ασχοληθεί με το ίδιο ακριβώς θέμα πριν από ένα χρονικό διάστημα. Θα ήθελα επίσης να πεθύνω θερμοχαιρετισμό και στον ε, Επίτροπο και να συγχαρώ τον εισηγητή και του συντάκτε ε, για την πολύ καλή δουλειά του. Όμως λυπούμε, Πρόεδρε, που είναι άδεια τα έδρανα του Συμβουλίου. Η ΕΤΕΠ είναι διοργανικό μέσον, ε, είναι δηλαδή εταίροι μέσα στην ΕΤΕΠ τα κράτη-μέλη τα ίδια. Ταυτόχρονα θα ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία που αποδίδουν και την τιμή ε, προ το Κοινοβούλιο, ο πρόεδρο Μεστάπ και όλο του το προσωπικό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερο. Η ΕΤΕΠ είναι μία τράπεζα η οποία ως εκ της εντολής της και της αποστολής της θα πρέπει να έχει και προληπτικό έλεγχο τον οποίο δεν έχει. Είναι μια διεθνή οργάνωση μη υπαγόμενη στους εθνικούς οργανισμούς ε, ελέγχου. Γι' αυτό λοιπόν ε, υποβάλλω τροπολογία έτσι ώστε η τραπεζική αρχή την οποία θέλουμε να θεσπίσουμε να έχει και μία περίμετρο ελέγχου προληπτικού ε, μέσα στις εντολές της. Και κύριε Επίτροπε θα ήθελα να εξηγήσω λίγο περισσότερο. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη αντιτίθενται σε αυτήν την πρόταση αλλά δεν μπορούν ε, οι στοδίνεκες να αναθέτουν εντολές ε, τα κράτη-μέλη και να μην επιτρέπουν το προληπτικό έλεγχο στην ΕΤΕΠ. Θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσω λίγο περισσότερο τι θέσει μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επενδύει αρκετά και το βλέπουμε αυτό. δεν πρόκειται για την διασύνδεση των μεταφορικών δικτύων, για τι ε, οδού μεγάλη ταχύτητα, για την εκπαίδευση, την υγεία, την ποιότητα των υδάτων. Χρειάζονται περισσότερε επενδύσει σε όλου αυτού του τομεί. Όμω, πολύ σωστά είπε ο πρόεδρο Μεστάτο ότι είναι ανεξάρτητη τράπεζα η ΕΤΕΠ και θα πρέπει να διατηρήσει τη διαβάθμιση τη στα τριπλό Α. Και άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο το 1-3 ευρώ. Αυτό είναι δυνατόν εφόσον όμως έχουμε έναν προϋπολογισμό επενδύσεων και, συνεργασία για τις, και συνεργασία για τις καινοτόμες επενδύσεις με την ΕΤΕΠ, κράτη-μέλη και ΕΤΕΠ. Αυτό νομίζω χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και αξιοποίηση του μέσου αυτού, του οργάνου αυτού που είναι τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών, για ένα λεπτό, το λόγο έχει ο κύριος Ιβάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ε, μια επιτυχημένη επιχείρηση, είναι τα πιο επιτυχημένα ευρωπαϊκά σχέδια και ακόμη και εν μέσω της κρίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατάφερε να, να διαφυλάξει την πιστοληπτική της διαβάθμιση των τριών α. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει πάντως να τύχει μια ριζικής επανεξέτασης της αποστολής της. Έχω τρία σχόλια κυρίως. Τα χορηγούμενα δάνεια θα πρέπει να συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020. Επίσης, τα δάνεια αυτά θα πρέπει να στηρίζουν ευρύτερα επενδυτικά προγράμματα για να μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να ανακάμψει πλήρως. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ε, πιο σταθερού και ισχυρού οικονομικού πλαισίου. Εκ μέρους των φιλελευθέρων και για δύο, λεπ... δυόμιση λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Μέστατ, κύριε Επίτροπε. Θα θέλω να ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ ενδιαφέρουσα και καλή έκθεση και να πω εκ μέρους της ε, ομάδας των φιλελευθέρων ότι συγχαίρουμε την ΕΤΕΠ για το εξαίρετο έργο της και την ταχύτατη αντίδραση την ώρα που μας έπληξε η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση. Απέδειξε δηλαδή η ΕΤΕΠ ότι είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις. Την ώρα που έπληξε την Ευρωπαϊκή Ένωση η οικονομική κρίση, η ΕΤΕΠ προέβη σε αύξηση κεφαλαίου ενίσχυση του δυναμικού της και έτσι μπόρεσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των καταστάσεων, στη βελτίωση των συνθήκων για όλους μας. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσω τη σημασία της ΕΤΕΠ και της αρρωγής που προσέφερε, γιατί χάρη σε αυτήν μπορέσαμε να ε, ελαφρύνουμε το άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι 90% των ε, επιχειρήσεων της Ευρώπης είναι μικρομεσαίες και ότι χάρη σε αυτές έχουν δουλειά 100 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε στις, ε, στις προσπάθειες της ΕΤΕΠ για την ανάπτυξη ε, μεταξύ άλλων και ενός δικτύου αποτελεσματικών, ενός διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεσματικών που χρειαζόμαστε εξάπαντος. Είδαμε άλλωστε τα διδάγματα από τις ε, συνέπειες της έκρηξης του ηφαιστείου της Ιρλανδίας. Χρειάζεται η ΕΤΕΠ να μας βοηθήσει και για την ε, πάταξη της διαφθοράς, πράγμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ομάδα μου. Και γι' αυτό ιδιαίτερω ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μα για το γεγονό ότι η ΕΤΕΠ ε, ακολούθησε τι πάγιε εδώ και μερικά χρόνια συστάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο ως προς τη διαφάνεια. Αποτελεί υπόδειγμα και για τα άλλα θεσμικά όργανα. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η ισότητα ευκαιριών μέσα στην ΕΤΕΠ δυστυχώ ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί αυτό είναι ένα αρνητικό, ένα μελανό σημείο στην ΕΤΕΠ. Πολύ λίγε είναι οι γυναίκε ε, μέσα στο προσωπικό τη ΕΤΕΠ, μόνο 20%. Κύριε Μίστατ, πρέπει να, δώσει, ε, να δώσει όθηση ώστε να αλλάξουν τα ποσοστά και οι αναλογίες αυτές μέσα στην ΕΤΕΠ. Πολύ καλή βαθμολογία λοιπόν εν γέννη, αλλά ένα, μία κοσμία ως προς την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ο κύριος Φιλίπ Λαμπέρεκ, μέρο των Πρασίνων. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μέιστατ, ε, κύριε συμπατριώτη, χρειαζόμαστε μια τράπεζα σαν την ΕΤΕΠ και μάλιστα έχουμε ανάγκη μια τέτοια τράπεζα όταν ε, οι ιδιωτικές τράπεζες ε, απέδειξαν ότι δεν επιτελούν την αποστολή της και απλώς ευλογούν τα γένια τους. Ουσιαστικά καταστρατηγούν το γενικό συμφέρον αντί να το εξυπηρετούν. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια τέτοια τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα πρέπει να λάβει αυξανόμενη σημασία και ισχύ. Και φυσικά ο ρόλο σα είναι καταλητικό. Μια τέτοια δημόσια τράπεζα σαν την ΕΤΕΠ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ε, τι ανάγκε τη αγορά ή να ανταποκριθεί σε όλε τι ανάγκε τη αγορά. Θα είναι καταλητικό ο ρόλο ρόλος σα όμω στη μεταμόρφωση των κοινωνιών και των οικονομιών μας για να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές προκλήσεις αυτών των χαλεπών καιρών και γιατί θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους περιορισμούς του πλανήτη, την εξάντληση των πόρων και τις κλιματικές αλλαγές, αλλά να ανταποκριθούμε και στην σημαντική αυτή πρόκληση της κοινωνικής συνοχής και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στον αναπτυξιακό κλάδο που είναι πολύ σημαντικός. Θα αναφερθώ σε ένα στοιχείο. Βλέπουμε τις επενδύσεις που χρηματοδοτείται στον ενεργειακό κλάδο και το 2009 τα τρία τέταρτα αφιερώνονταν σε τεχνολογίες του 19ου και 20ου αιώνα και μόνο ένα τέταρτο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε η πρόκληση για την ΕΤΕΠ είναι να αντιστρέψει αυτές τις αναλογίες. Δηλαδή από το 2010 και μετά τα τρία τέταρτα των επενδύσεών σας και των συνολικών δανείων ε, να χρηματοδοτούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες. Και εκεί είναι που θα διαδραματίσετε τον καταλητικό σας ρόλο, γιατί θέλουμε πραγματικά να γίνει πρώτη τάξη ως τράπεζα σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Για ένα λεπτό το λόγο κύριο Τσαρνέτσκι. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας, τον κύριο Ταμάς Ντόιτς, για την πολύ αξιόλογη του έκθεση και νομίζω ότι η αύξηση του όγκου ε, που ζητά για την ΕΤΕΠ η έκθεση είναι πολύ φιλόδοξη. Τώρα για τον Ευρωπαίο ψηφοφόρο και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί χρηματοδοτεί κυρίως ε, προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Γι' αυτό και είμαστε υπέρ της αύξησης του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και της ενίσχυσης των δανείων που χορηγεί. Γιατί η ΕΤΕΠ υποστηρίζει ένα τομέα που έχει ανεκτήμητη σημασία για τον Ευρωπαίο πολίτη, που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εγώ ως Πολωνός θα ήθελα να πω ότι ελπίζω ότι η ΕΤΕΠ θα στηρίξει τη μεταμόρφωση και στη δική μας περιοχή της Ευρώπης με σημαντική συμβολή. Ήδη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, έχει αναλάβει σημαντικές ε, δεσμεύσεις και για μας έχει άμεση σημασία αυτή η ανάμειξη της Τράπεζας Επενδύσεων και στην περιοχή μας. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρώπης Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Ανδρέασεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν κοιτάω τι προγράμματα χρηματοδοτεί η ΕΤΕΠ, βλέπω ότι υπάρχουν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και αναρωτιέμαι πώς θα βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. General Motors, Electrogroups, Arsenal Metal χρειάζονται την ΕΤΕΠ και τους ήπιου όρου που προσφέρει. Σε τι βοηθούν αυτά τα δάνεια. Δημιούργησαν νέε θέσει εργασίας. Όχι, εξήγαγαν θέσει εργασία χάσαμε θέσει εργασία από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Electrolux, για παράδειγμα, είναι παράδειγμα επιτυχία τη ΕΤΕΠ. 250 εκατομμύρια για να ενισχυθούν οι δυνατότητε τη επιχειρήση με νέα εργοστάσια στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και αλλού. Και όταν τελείωσε εκεί η παραγωγή, χάθηκαν 2.000 θέσει απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για το ότι η ΕΤΕΠ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδιαίτερα στο ισοζύγιο εμπορίου, διότι χάνονται θέσεις απασχόλησης και αυξάνεται η ενέργεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων για ένα λεπτό ο κύριος Χανς Πέτερ Μάρτεν. Α, όχι, δεν είναι εδώ. Οπότε ο κύριος Μέλτσερ μου λένε ότι έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ κύριε Μέλτσερ. Ευχαριστώ πρόεδρε βλέπουμε από την ετήσια έκθεση ότι, έχουν, ε, ότι αντέδρασε γρήγορα η ΕΤΕΠ ε, στην, κρίση, στην οικονομική κρίση με προτεραιότητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανάπτυξη του δυναμικού της περαιτέρω. Πλην όμως θα πρέπει να δούμε αν όντως έφτασαν στις ε, μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις τα δάνεια, οι πιστώσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλό να ιδρυθεί μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας των Τραπεζών με αποτελεσματική δουλειά, με αποτελέσματα ουσιαστικά και ε, αυτό προϋποθέτει σημαντικές αρμοδιότητες και την δυνατότητα να ελέγχει, να υποπτεύει υπερσυνοριακά εργαζόμενες τράπεζες. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε περισσότερο να ε, στήσουμε στην, ε, στις δραστηριότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντοπιστούν οι δυσκολίες, τα προβλήματα όπου υπάρχουν και να μην ε, βλέπουμε επανάληψη ή επικάλυψη εργασιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ και με αυτές τις παρεμβάσεις. Τελειώνουν οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων των ε, πολιτικών ομάδων που μιλάνε εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και περνάμε τώρα στον γύρο μιλητών που μιλούν σε προσωπικό επίπεδο. Για 1,5 λεπτό πρώτο ο κύριος Σον Κέλλη. Πρόεδρε, συμφωνώ με τους συναδέλφους που μίλησαν με εγκομιαστικά λόγια για την ΕΤΕΠ. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και τι είδους ε, παιχνίδια έχουν επεχθεί με τις ε, ιδιωτικές τράπεζες, με τα μεγάλα πακέτα ε, επιχορηγήσεων, τα μπόνους και τον, την ανεξέλεκτη δραστηριότητά τους. Η ΕΤΕΠ, ίσως επειδή λέει ο Πρόεδρος έρχεται να λογοδοτήσει το Κοινοβούλιο, πρέπει να επενεθεί αντίθετα από τις άλλες τράπεζες για τις δραστηριότητες της και ιδιαίτερα την πέμπτη δράση και την ε, ε, βοήθεια που προσέφερε μέσα στην οικονομική κρίση. Ιδιαίτερα δε επειδή δίνει υποστήριξη και αρρωγή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 300 εκατομμύρια χορηγήθηκαν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την ΕΤΕΠ στη δική μου την πατρίδα, την Ιρλανδία. Όμως το, το θέμα που τίθεται είναι αν όντω φτάνουν μέχρι τι μικρομεσαίες επιχειρήσει τα χρήματα αυτά και αν όχι γιατί και γιατί απορρίπτονται κάποιε αιτήσει δανείων από επιχειρήσεις οι οποίες όμως έχουν καλό επιχειρησιακό σχέδιο. Όταν ορισμένε επιχειρήσεις βλέπουμε να, να χρεοκοπούν στην Ιρλανδία ιδιαίτερος ε, ενώ υπάρχουν χρήματα προς διάθεση, βλέπουμε ότι δεν έχουμε βγει ακόμη από την κρίση. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι απορροφούν ε, οι ιδιωτικές τράπεζες κονδύλια τα οποία θα πρέπει να απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για άλλες δικές τους δραστηριότητες. Αληθεύει αυτό, γιατί έτσι ακούγεται. Και εάν ναι, πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτά τα περιστατικά. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γκάιερ. Πρόεδρε, κύριε Μαρτίνες, πρόεδρε, κύριε Μάιστατ, κύριε Επίτροπε Ρεν, θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον ε, κύριο Ντόιτ, τον συνάδελφο, για τη δουλειά του και ταυτόχρονα να ε, εξάρω τη σημασία τη ΕΤΕΠ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολίτε τη Ευρώπη. Μέσα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης όπως η σημερινή βλέπουμε τι σημασία έχει η ΕΤΕΠ ως μέσο αντιμετώπισης κρίσης. Βεβαίως, και η ενίσχυση της αποδοτικότητας ε, των προγραμμάτων όπως ε, κρίνεται άλλωστε με τους ελέγχους, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ αξιόπιστη η ΕΤΕΠ, ότι μπορεί με, τις, με τα έξι ενδοτικά της προγράμματα να στηρίξει τα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να βοηθήσει γενικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης και την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε. Ταυτόχρονα βέβαια ως Ευρωβουλευτές πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω το δυναμικό της, ιδιαίτερα τα επενδυτικά της μέσα. Και για την ομάδα μου μεγάλη σημασία έχει το αίτημα που θέλουμε να απευθύνουμε στην ΕΤΕΠ, ότι δηλαδή ε, βεβαίως θα πρέπει να εξετάζει τα θέματα των εξωχωρίων ε, ε, επενδύσεων, χωρίς όμως να επιτρέπει την διαρροή χρημάτων σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Για ένα λεπτό τώρα, συνάδελφος Γουρίνς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι συγχρόνως και τράπεζα και θεσμός όργανο. Και ως τράπεζα δεν μπορεί να ξεχάσει ότι είναι θεσμός και όργανο και ως θεσμός και όργανο δεν μπορεί να ξεχνάει ότι είναι και τράπεζα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αγνοεί την επαναχρηματοδότηση που πρέπει να προσφέρει. Δεν πρέπει να μπαίνει σε άχρηστου κινδύνους, ιδιαίτερα με επενδύσει σε υπονάπτυξη χώρε. Είναι πολύ σημαντικό όμω να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου στους θεσμικούς δανειστές ε, να μπορούν να παρεμβαίνουν ως δωρητές, ενώ η ΕΤΕΠ να κάνει δάνεια. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι έγινε με την Παγκόσμια Τράπεζα η οποία αναγκάστηκε να ακυρώσει δισεκατομμύρια χρεών επειδή δεν εξοφλήθηκαν. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή στις δράσεις της ΕΤΕΠ, η οποία ελπίζω να μπορέσει να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητες της στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ευχαριστούμε κύριε Γούρενς. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Μπεναβαγατού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην έκθεσή σας του 2008 επιμένετε οι εξωτερικές δραστηριότητες της τράπεζας να είναι σύμφωνες με τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό και το σχέδιο χρηματοδότησης πυρηνικών σταθμών είναι κάτι που αντιβαίνει στο άρθρο 3, παράγραφος 5 της Εθήκης της Ένωσης που λέει ότι στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην αηφόρο ανάπτυξη του πλανήτη. Το Φεβρουάριο του 2009 οι αρχές της Ιορδανίας λοιπόν ήρθαν σε επαφή με την ΕΤΕΠ για να ζητήσουν στήριξη ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας εκεί, ιδιαίτερα με την οικοδόμηση πυρηνικού σταθμού. Με ικανοποίηση λοιπόν λοιπόν η υπηρεσία σα με... πήρε τη διαβεβαίωση από την υπηρεσία σα ότι η ΕΤΕΠ δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημα αυτό και ότι θεωρεί πώ πρέπει να στηρίζει αναπτυξιακά προγράμματα για την αιωλική ενέργεια και ηλιακή ενέργεια στην Ιορδανία, που είναι και η ενέργεια του μέλλοντος για την ανανεώσιμη πηγή ενέργεια ε, ο ήλιο και αέρας. Ελπίζω να γίνει το ίδιο και για άλλε αιτήσει που λαμβάνετε που θα λάβετε για στήριξη στην πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Για ένα λεπτό τώρα, ο Κόβαλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η σταθερότητα της Ουκρανίας είναι βασικός στόχος για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για χώρα που αποτελεί εταίρο μας. Ξέρουμε ότι περνάει από κρίση η χώρα, η Ουκρανία και η σταθερότητα στη χώρα αυτή είναι πολύ βασική και για την οικονομική της σταθερότητα. Η πολιτική της δηλαδή είναι σημαντική για την οικονομική της σταθερότητα. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε αυτή τη χώρα, γιατί όσο πιο πολύ την στηρίζουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να έχει μεταρρυθμίσεις η χώρα αυτή που θα την κάνει να περάσει στην οικονομία αγοράς. Και η κρίση της Ουκρανίας δεν είναι κρίση μόνο της Ουκρανίας, είναι και δικό μας πρόβλημα. Γιατί σήμερα περνάμε από μια δοκιμή. Σε τι βαθμό είμαστε σε θέση, μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα. Εγώ είμαι υπέρ της μακροοικονομικής ενίσχυσης στην Ουκρανία λοιπόν και ήρθε η ώρα σήμερα να πούμε ότι η ενίσχυση αυτή πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο γιατί έτσι και οι προσδοκίες μας από τη χώρα αυτή μπορούν να είναι ακόμα μεγαλύτερε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόβαλ. Τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ο συνάδελφος Αλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι επιτυχή στα 52 χρόνια της λειτουργίας της ιδιαίτερα στην επίτευξη και ενίσχυση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τον κορμό των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούν τον κορμό των επιχειρήσεων εκείνων που πρέπει να διατηρηθούν στα πλαίσια της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και εντεύθυν την κοινωνική ηρεμία στην Ένωση. Σήμερα βέβαια είναι γνωστό ότι η Ένωση αντιμετωπίζει την ελληνική κρίση. Δεν γνωρίζω βέβαια εάν ο ιστορικός του μέλλοντος θα την ονομάσει η ελληνική κρίση ή η οικονομική κρίση ή ίσως την ονομάσει και νομισματική κρίση. Να το δούμε αυτό. σίγουρα γνωρίζω ότι ο Γαλιλαίος εάν ζούσε σήμερα δεν θα έλεγε ότι η γη γυρίζει, θα έλεγε η γη τρέχει. Διότι τρέχουν πολλά γεγονότα τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δώσουμε τις απαραίτητες λύσεις. Ε, θεωρώ ότι όλοι εδώ μέσα πιστεύουμε ότι ο ομαλός βίος της Ένωσης επιβάλλει την επιτάχυνση στην ολοκλήρωση της πολιτικής και της οικονομικής της ενοποίησης. Στα πλαίσια αυτά θεωρώ ότι η ΕΤΕΠ έχει την τεχνογνωσία και την αντικειμενική δυνατότητα να αναλάβει και άλλες δράσεις και προτείνω να εξεταστεί ιδιαίτερα το προτείνω στον κύριο Όλι Ρεν ε, στην σοβαρότητα του οποίου έχω μεγάλη εκτίμηση να εξετάσει το ενδεχόμενο του ρόλου της ΕΤΕΠ μελλοντικά ίσως στο ρόλο του ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών μελών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό τώρα. Το λόγο έχει ο κύριος Μάρτιν. Βεβαίω. Ήδη επεσήμαναν, Πρόεδρε, οι συνάδελφοι τη σημασία της ΕΤΕΠ. Η κυρία Κάρνμπαχ μίλησε ε, για την ανάγκη να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Εγώ θα ήθελα όλα αυτά να τα θέσω σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε α, κράτη, σε κράτη πολλά να επικρατούν τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και γιατί δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή όπως αντιθέλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε αυτές, ε, ε, αυτή η άκρα δεξιά να συγκαλύπτεται κάτω από το μανδύα του προβάτου, του αμνού. Γιατί βλέπουμε να ε, βάλουν κατά δικαίων και αδίκων. Εμένα πρόσφατα κάποιοι τέτοιοι με απεκάλεσαν ψυχοπαθή. Αυτή είναι η ορολογία του Χίτλερ, αυτή είναι η ορολογία του φασισμού και παρακαλώ και τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσουν τη δουλειά τους και με όρους διαφάνειας. Όσο πιο διαφανείς είναι οι όροι με τους οποίους μιλάμε, τόσο πιο εύκολο θα μπορέσουμε να πατάξουμε τον νεοφασισμό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σοφία Κονή για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Με την έκθεση για το 2008 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων γιορτάζουμε μια επέτειο. Πέρασαν πάνω από 50 χρόνια που η ΕΤΕΠ συμβάλλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επίρου. Γιατί με μακροπρόθεσμα δάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Επίσης χαίρομαι για τις νέες ρυθμίσεις από τον ε, φθινόπωρο του 2008. Μέσα σε μία χρονιά μόνο πρόσθεσε 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις προβλέψεις της και ως μέλος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και τα δάνειά της προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να ε, να χρηματοδοτούμε πρωτοβουλίες όπως το Τζέρεμι γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται τεχνική αρρωγή, ε, ίδια κεφάλαια, δάνεια σαν αυτά που προβλέπει το Τζέρεμι. Και μάλιστα στην περιφέρεια της Οβέρνη εδώ και ένα χρόνο έχουμε ένα ειδικό μηχανισμό ενίσχυσης προς τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 25 εκατομμύρια ευρώ, 18 από το ΦΕΝΤΕΡ που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να εξέλθουν από την κρίση χρησιμοποιώντας τις καινοτόμες τεχνολογίες. Χαίρομαι για, τις, ε, για την πολύ αγαστή συνεργασία της ΕΤΕΠ, του Αναπτυξιακού Ταμείου και των τοπικών και περιφερειακών αρχών και σας ενθαρρύνω κύριε Μέιστατ να συνεχίσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε κύριο Οκονή. Για ένα λεπτό Τάις, ο κύριος Τάις Μπέρμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ΕΤΕΠ έδρασε πολύ σωστά και ανταποκρίθηκε με την ε, αύξηση του κεφαλαίου της και διπλασιασμό των επενδύσεων και των δανείων ιδιαίτερα προς οι μισές επιχειρήσεις ε, σε σχέση με πέρυσι. Στις εξωτερικές, ε, στην εξωτερική εντολή όμως δεν είχαμε εντυπωσιακέ αλλαγέ προ τι ε, αναπτυσσόμενε χώρε. Και μάλιστα στι χώρε ΑΚΕ, στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, μειώθηκαν τα δάνεια τη ΕΤΕΠ. Και μάλιστα και στι αναπτυσσόμενε χώρε ε, ήταν πολύ βραδύτερη η αντίδραση της ΕΤΕΠ. Είναι δημόσιος οργανισμός η ΕΤΕΠ, οπότε δεν θα πρέπει να επενδύει μόνο σε βαριές υποδομές της αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα άλλο σημαντικό της έργο είναι να προσφέρει κεφάλαιο σε περιοχές ε, ισχνών αγελάδων και μάλιστα εκεί που είναι απρόθυμες ιδιωτικές τράπεζες. Θα πρέπει Επίση, να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση σε αποταμιεύσει και δάνεια και για πολίτες και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε αηφόρο ανάπτυξη, όχι μόνο εδώ, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σα ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, το λόγο έχει ο κύριο Σταυρακάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πριν καλωσορίσω στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον πρόεδρο maystadt και τον συγχαρώ τόσο για τις επιτυχημένες δραστηριότητες της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων όσο και το φιλόδοξο επιχειρησιακό της σχέδιο θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη μου για την εμπριστική δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν στην αθήνα χθε τρει συμπολίτε μου στον χώρο εργασία του και να εκφράσω επίση τα ειλικρινά μου σε συλληπιτήρια στι οικογένειέ του δεν υπάρχει αμφιβολία κύριε πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι η σημερινή οικονομική κρίση ανέδειξε και το σημαντικό έργο της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων. η πρόσθετη χρηματοπιστωτική υποστήριξη της ετεπ επέτρεψε γρήγορε εκταμιεύσει και συνέβαλε στην στήριξη τη πραγματική οικονομία ιδίω προστατεύοντα τα ωφέλιμα έργα και βοηθώντα τι βιώσιμε επιχειρήσει σε αυτού του εξαιρετικά δύσκολου καιρού. επίση σημαντικό κομβικό ήταν ο ρόλο τη ετεπ στο κεντρικό πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, όπου με τη μορφή Jaspers και Jeremy η ΕΤΕΠ προώθησε ακόμη περισσότερα εργαλεία για να συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη της καινοτομίας. Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος της ΕΤΕΠ αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο στο πλαίσιο των στόχων συνοχής αλλά και στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μέσω των ευφυών εργαλείων χρηματοοικονομικής μηχανικής που αναπτύσσει διαρκώς με, την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία Έλενα, Ευρωπαϊκή Τοπική Βοήθεια για την Ενέργεια, αναμένεται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω αξιόλογων επενδύσεων σε τομείς όπως η αηφορία, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σα ευχαριστούμε κύριε Σταυρακάκη. Το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια δρυμύτατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε όλους μας και μάλιστα η υποστήριξη της ΕΤΕΠ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αύξησε κατά 42% τη χορήγηση δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητά τους για την ευρωπαϊκή οικονομία. Συνεχίζεται δυστυχώς η χρηματοπιστωτική κρίση, καλπάζει η ανεργία και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε διατήρηση και συνέχιση της ε, υποστήριξης ΕΤΕ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ξεπεράσουν ε, τα προβλήματα ρευστότητας ε, και χαμηλής πρόσβασης που έχουν στο κεφάλαιο. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτιμήθηκε ιδιαίτερα στις χώρες που επλήγησαν δρυμύτερα από την κρίση και πιστεύω ότι η τράπεζα αυτή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε σχέδια υποδομών, ενέργειας και μεταφορών. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο ο κύριος Πρόεδρο Δερόσα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σήμερα θα προσπαθήσαμε απεγνωσμένα να την ιδρύσουμε. Χαίρομαι για την πρόταση αύξησης, ενίσχυσης του όγκου των δανείων και την παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μερικές φορές όμως διασπαθεί με αυτό τον ανεκτήμητο πόρο γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε αρκετά την εμπειρογνωμοσύνη του. Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι σοσιαλιστέ προτείνουν την ίδρυση ενό trust fund. Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να πατάξουμε την ανελαιή επίθεση, επίθεση των ε, κερδοσκόπων και θα εξασφαλίσουμε χαμηλότερα spread. Έτσι θα δείξουμε στην αγορά και στους κερδοσκόπους ότι δεν θα επιτρέψουμε την καταβαράθρωση κανενός κράτου και την καταστροφή κανενός κράτου όπως συμβαίνει σήμερα στην ε, Ελλάδα και πολύ πιθανό να συμβεί ε, στο μέλλον και με άλλες χώρες, ίσως και με τη δική μου πατρίδα την Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ και η τελευταία ομιλήτρια στη συζήτηση αυτή πριν να περάσουμε στο Catch the Eye και για ένα λεπτό το λόγο κυρία Κορίνα Κρέτσου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο πλαίσιο της κρίσης ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, αντέδρασε άμεσα, τροποποίησε τις προτεραιότητές της και αύξησε τη χορήγηση δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι αυτές που εκτέθηκαν πολύ περισσότερο στη χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει να δούμε όμως ε, πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξασφαλίσει τη συγχρηματοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων στις νέες χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους ε, και στις ε, τοπικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις κεφαλαίες Οι νεότερες αυτές χώρες της Ένωσης δεν καταφέρουν να, να δώσουν όθηση στην οικονομία τους και να αποφύγουν ε, την οικονομική και κοινωνική παρακμή. Χρειαζόμαστε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την οικονομική ανάκαμψη και στις χώρες αυτές και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και έχει πια νομική προσωπικότητα, να καταστεί μέτοχος της τράπεζας και να ενισχύσει το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και της συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε κυρία Κρέτσου. Περνούμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye, αλλά για μισό λεπτό προηγουμένως ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μέλτσερ γιατί κάποιος συνάδελφος έκανε προσωπικό υπενημό προς τον κύριο Μέλτσερ. Πρόεδρε, επικαλούμε το άρθρο 150 του κανονισμού για μια, προφο... μια προσωπική παρατήρηση. Ο Χάνς Πέτερ Μάρτεν ε, στην ομιλία του εξέπεμψε ε, σημαντικές κατηγορίες εις βάρος του μου και νομίζω ότι εκείνος ο βουλευτής ο οποίος έχει κάνει επάγγελμα τις ε, καταγγελίες εις βάρος συναδέλφων του μέσα από τον τύπο και εκείνος ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει μεθόδους ε, μυστικών υπηρεσιών με κρυφές κάμερες, με μικρόφωνα κρυμμένα στο πέτο. Δεν μπορεί να μιλήσει για κανέναν άλλον. Δεν, έχω ποτέ, δεν είχα ποτέ και δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Δεν του έχω ποτέ απευθύνει το λόγο και γι' αυτό απορρίπτω με τα στις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τις αποσύρει. Ευχαριστώ για τα λόγια σας. Το λαμβάνουμε υπόψη μας. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye. Έχουμε πέντε συναδέλφους που έχουν ε, ζητήσει το λόγο σύμφωνα με τον κανονισμό. Ο κύριος Λουκαν Πέτου πρώτα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ΕΤΕΠ για τις προσπάθειές της προκειμένου να πετύχει τους κοινοτικού στόχους. Έχει σημαντικό ρόλο να παίξει η ΕΤΕΠ, ιδιαίτερα μέσα σε μια περίοδο κρίσης, ζωτικής σημασίας. Ο στόχος της σύγκλησης πρώτα απ' όλα. Οι σχετικές περιφέρειες παίρνουν χρήματα και από το Ταμείο Συνοχής και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Βασικός στόχος της τράπεζας, 28 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 41% των πιστώσεων της ΕΤΕ πάνε σε προγράμματα τα οποία εγγράφονται ακριβώς σε αυτά τα πλαίσια. Πιστεύω όμως ότι οι πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης ε, δεν μπορούν να βοηθηθούν παρά μόνο εφόσον διαθέτουν υποδομές για την κατάρτιση, κοινωνικές υποδομές που να ανταποκρίνονται όμως τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Γι' αυτό λοιπόν ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει τις δράσεις της για να προωθήσει την κοινωνική συνοχή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζορτ ε, Πούτες. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει να παίξει βασικό ρόλο για να ενισχυθεί η σύγκληση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα σε περίοδο κρίσης όπου πρέπει να γίνονται επενδύσεις από το δημόσιο τομέα. Η ΕΤΕΠ κατά την περίοδο κρίση ανταποκρίθηκε με ταχύτητα και η Ρωμανία πήρε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕΤΕΠ μέσα στο 2009. Κάτι το οποίο δείχνει με ποιο τρόπο η τράπεζα συμμετέχει στι προσπάθειες για να ε, περιοριστούν ε, οι ζημιές ε, από την κρίση μετά την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσβαση σε κεφάλαια επίσης από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται αυτό και να έχουμε πιστώσεις που δίνονται με διαφάνεια για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Αντρικένη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, μάλιστα, κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να υπογραμμίσω και να εξάρω τον πολύ σημαντικό ρόλο τη ΕΤΕΠ στην ε, ανάταξη και ανοικοδόμηση των οικονομιών μα, ιδιαίτερα στι δύσκολε περιστάσει που γνωρίζουμε. Η πατρίδα μου, η Λιθουανία, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στην οποία η ΕΤΕΠ έχει προσφέρει με τα μέτρα για την ανάταξη της οικονομίας, ε, για την διέξοδο από την κρίση, για τη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προγραμμάτων μεταφορών και θα ήθελα να ε, ε, παρακαλέσω τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προσφέρουν περισσότερο δυναμικό και, στις, ε, και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιπλέον έτσι ώστε να βοηθήσει και τις άλλες χώρες, ιδιαίτερα τις, ε, τους γείτονες μας τα ανατολικά με τις ενισχύσεις που ε, χρειάζονται για επενδύσεις, ιδιαίτερα στις μεταφορές, στο περιβάλλον αλλά και πάνω απ' όλα στην ενέργεια. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα τον τομέα της ενέργειας γνωρίζοντας πόσα προβλήματα στις υποδομές ενέργειας έχουν τα κράτη αυτά. Το λόγο έχει ο Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να ενώσω τη φωνή μου στα εγκόμια προς την ΕΤΕΠ και στα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και να συγχαρώ επίσης και τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντόιτς. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να διακρίνουμε στη συζήτηση δύο στόχους, ε, αφενός την ανάπτυξη και αφετέρου τη σταθερότητα, τη σταθεροποίηση. Με αυτή τη σειρά. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να συμβάλλει προς τη συνοχή. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο τη ΕΤΕΠ για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το είδαμε και στην περίπτωση της ε, Λισαβόνας ότι χωρίς ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χωρίς περιφερειακή συνεργασία δεν θα τα καταφέρουμε. Επίσης, ε, οι γειτονικέ χώρες ε, της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης χωρίς την βοήθεια και τη συμβολή της ΕΤΕΠ δεν θα καταφέρουν να, να ορθοποδήσουν. Δυστυχώς διακόπτει το μικρόφωνο ο κύριος Μαρτίνης, το λόγο ο κύριος Ρούμπιχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Μάιστατ, θα ήθελα να μου πείτε πώς προχωρούν τα πράγματα σχετικά με τη συζήτηση ως προς την Βασιλεία Τρία, τι πρόοδος υπάρχει, τι τάσεις διαγράφονται και σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Πιστεύετε λοιπόν ότι εδώ μπορούμε να ε, περιμένουμε θετικές εξελίξεις ως προς ε, τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για να διεξέλθουμε από την κρίση ή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμη και επίσης ε, τι είδους δυνατότητες έχουμε για ενίσχυση των επιχειρηματικών και των επιχειρησιακών κεφαλαίων, κεφαλαίων κινδύνου που χρειάζονται να διατεθούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων το τι θα μας πείτε και ευχαριστώ ιδιαίτερος ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την πολύ καλή συνεργασία και με την ΕΤΑ και την υποστήριξη προσφέρει μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφενός αλλά και τα, διεθνή, ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα αφετέρου. Ευχαριστώ πολύ και με την παρέμβαση του κυρίου Ρούμπιχ τελειώνει ο γύρος του Catch the Eye. Όχι, όχι. Το λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος Μάιστατ για να σχολιάσει όλα αυτά που άκουσε από τους προλαλήσατες στη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους παρενέβησαν στη συζήτηση για τις παρατηρήσεις τους και σίγουρα πολλές ερωτήσεις χρήζουν ευρυθέστερης και εκτενέστερης συζήτησης εγώ ακροθυγώ θα δώσω κάποιε απαντήσει. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τι επιχειρησιακέ μα προτεραιότητε, θα ήθελα να πω δύο λόγια και επίση να μιλήσω λίγο για τον έλεγχο τη διακυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τι επιχειρησιακέ μα προτεραιότητε, μία από αυτέ ε, επισημάνθηκε από πολλού ομιλητέ ε, που αναφέρθηκαν στην υποστήριξη που χρήζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυρία Γκιόρη, για παράδειγμα, και ο κύριο Σμίτ αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα αυτό και σωστά επιμένουν στην ανάγκη υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 2008 φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πως εγκαινιάσαμε ένα νέο προϊόν για τα δάνεια προς τις τράπεζες που θα, χρηματοδοτήσουν τις, ε, θα δανειοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να παρακολουθήσουμε καλύτερα την ε, αξιοποίηση και τη χρήση των ε, δανείων που χορηγούμε. Το πρώτο τρίμηνο του 2008 και μέχρι τα τέλη του 2009 ε, υπογράψαμε δάνεια 21 δις. 16 δις ήδη έχουν ε, ε, χορηγηθεί και πάνω από 90% των ποσών αυτών πέρυσι είχαν όντως χορηγήσει δάνεια είχαν δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τις εμπορικές τράπεζες και παρακολουθούμε την χρήση αυτών των κονδυλίων και όπως είπε και η κυρία Γκιορή, επιλέγουμε ως ενδιάμεσους ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όχι μόνο τις εμπορικές τράπεζες αλλά και τις εμπορικές τράπεζες και τα ταμιευτήρια και έχουμε πολύ ε, ευρύτερο φάσμα πλέον ενδιάμεσων ε, εταίρων. Επίσης διαλέξαμε και κάποιες συνδυασμένες δραστηριότητες και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα δώσει εγγύσεις στα χαρτοφυλάκια δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η κυρία Κονή αναφέρθηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα τέτοιες ε, συμμετοχής και συνεργασίες και σας ευχαριστώ θερμά για τα θερμά σας λόγια υποστήριξης προς την ΕΤΕΠ. Δεύτερη επιχειρησιακή προτεραιότητα της ΕΤΕΠ που αναφέρατε είναι το θέμα της σύγκλησης σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσπαθεί να ενισχύσει τις ενέργειες, τις δραστηριότητες της, τις περιφέρειες της σύγκλησης και μάλιστα το 2009 ο όγκος των δανείων μας αυξήθηκε περισσότερο στις νέες χώρες μέλη, στις τελευταίες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε τη βούληση να συμβάλλουμε στη μείωση του χάσματος και των διαφορών μεταξύ των χωρών μελών. Αυτή είναι και η τη της σύγκλησης άλλωστε. Και υπό αυτό το πρίσμα, όπως ε, επισήμαναν η κυρία Κάντερμπαχ και ο κύριος Τσαρνέτσκι, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση των διαρθρωτικών κονδυλίων. Και αυτό συμβαίνει. Αποκινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε διάφορα προγράμματα. Το Jaspers για την τεχνική αρρωγή για την προετοιμασία σχεδίου για να υποφεληθεί κανείς από τα διαρθρωτικά ταμεία. Την πρωτοβουλία Jeremy που μετατρέπει ουσιαστικά τα διαρθρωτικά ταμεία σε χρηματοπιστωτικό μηχανισμό με ένα χαρακτήρα revolving, τη δυνατότητα δηλαδή πολλαπλής χρησιμοποίησης του ίδιου ποσού και την πρωτοβουλία Jessica που επίσης χρησιμοποιεί τα διαρθρωτικά κονδύλια για καινοτόμε πρωτοβουλίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τρίτη επιχειρησιακή μα προτεραιότητα είναι η ενέργεια και η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και ίσω θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε πιο διεξοδική συζήτηση για το θέμα αυτό. Πάντω, σίγουρα συνιστά αυτό επιχειρησιακή μας προτεραιότητα και μαζί με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κ. Λάμπερτς μίλησε για την περίοδο 2002-2008 και μας ανέφερε εκεί τα αριθμητικά στοιχεία. Θα δείτε όμως ότι ήδη το 2009 αρχίζει και ανατρέπεται αυτή η τάση γιατί το 2009 Αφιερώσαμε πάνω από 4 δισεκατομμύρια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή 70% της χρηματοδότησης για την ε, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε αυτή η αντιστροφή των τάσεων συνεχίζεται υπέρ ε, μεγαλύτερης χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εδώ τον κύριο Σταυρακάκη που αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Έλενα, κοινό πάλι πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή τεχνική αρρωγή σε θέματα ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα και πάλι για την ενέργεια να πω στην κυρία Μπεναράμπα του ότι σεβόμαστε τις επιλογές των κρατών μελών για το μείγμα των πολιτικών, το policy mix. Αν μια χώρα επιλέξει την πυρηνική ενέργεια, δεν θα την αποτρέψουμε εμείς. Στην περίπτωση της Ιορδανίας όμως, εξετάζουμε μόνο προγράμματα χρηματοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δύο λόγια για τον έλεγχο τώρα και τη διακυβέρνηση. Ο κύριο Σοντή γνωρίζει τη θέση μα για την εποπτεία. Είμαστε διαλλακτικοί και ανοιχτοί. Ούτω ή άλλω ε, ελεγχόμαστε από μια ανεξάρτητη επιτροπή επιτήρηση, από το ελεγκτικό συνέδριο για τα χρήματα που λαμβάνουμε από τον κοινοτικό προπολογισμό. Ελεγχόμαστε από την Όλαφ, από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι είμαστε η διεθνή χρηματοπιστωτική οργάνωση που ελέγχεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Αλλά χρειάζεται και ίσως και, και μια τραπεζική εποπτεία και γι' αυτό είμαστε διαλλακτικοί και ανοιχτοί προς οποιαδήποτε πρόταση που θα υποβληθεί μέσω της νέας ε, Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής Εποπτείας. Για την, το τρίτο πακέτο της Βασιλείας παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στις ε, εργασίες, αλλά βρισκόμαστε ακόμη σε φάση διαβούλευσης για τη Βασιλεία 3, οπότε δεν έχουν αποκρισταλωθεί όλες οι παράμετροι. Σε ό,τι αφορά τα εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα, τα offshore, χρηματοπιστωτικά κέντρα. Σίγουρα αυτό το θέμα μας απασχολεί ιδιαίτερα και θα ήθελα να μπορούσα να σας δώσω περισσότερες διευκρινήσεις για τη νέα πολιτική της ΕΤΕΠ. Σίγουρα θέλουμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και την, τις φορολογικούς παραδείσους ή τη χρήση των εξωχώριων κέντρων για την φόρο αποφυγή. Και επίσης θα ήθελα να πω στον κύριο Σμιτ ότι δίκιο έχει, ότι έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο να διονύσουμε και να εξασφαλίσουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών, ιδιαίτερα στα στελέχη της, ανώτερα στελέχη της ΕΤΕΠ. Μάλιστα εγκρίναμε ένα νέο σχέδιο δράσης ε, που ε, πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να διορθώσουμε αυτή την έλλειψη στο μέλλον. Πάντως, ε, όντως, η σημερινή κατάσταση είναι απαράδεκτη ως προς την ισότητα των δύο φύλων στην ΕΤΕΠ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος Όλη Ρεν για να αντιδράσει στις παρεμβάσεις των ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την τόσο επικοδομητική συζήτηση που μπορέσαμε να έχουμε εδώ σήμερα. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάιτς για την εξαίρετη εκθεσή του. Επιπλέον, θέλω να πω τρία πράγματα. Πρώτον, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ότι η συζήτηση αυτή και η έκθεση αυτή θα δημιουργήσουν ένα εξαίρετο σημείο κίνησης για το μέλλον. Μπορούμε τώρα πολύ γρήγορα να προχωρήσουμε στην έγκριση της, εξωτερικής, της νέας εξωτερικής εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους εξωτερικούς μας στόχους, ιδιαίτερα την αναπτυξιακή μας πολιτική. Επιπλέον, Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό εταίρο που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη της στρατηγικής 2020 και κυρίως την εφαρμογή της, αηφόρος ανάπτυξη και απασχόληση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η σχέση αυτή. Επίσης, η ΕΤΕΠ μπορεί να δημιουργήσει δομές που στηρίζουν τις επενδύσεις και στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και συνεργαζόμαστε στενά μεταξύ μας. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Το τρίτο μου σημείο είναι το εξή. Πολλοί από εσά ανηφέρθηκαν στην ε, κρίση στην Ελλάδα. Ειλικρινά, χτες ήδη στην συζήτηση που έγινε εδώ εξέφρασα την θλίψη μου για τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους αιτίας βίων διαδηλώσεων χτες στην Αθήνα. Η δημοκρατία έχει το δικαίωμα να εκφράζεται, αλλά ποτέ με τη βία. Κάπου πρέπει να μπει το όριο. Και το όριο αυτό είναι ακριβώς η βία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να σταθεροποιήσει την ελληνική οικονομία. Σχεδιάζουμε και σχεδιάσαμε ένα μεγάλο πακέτο υπέρ της Ελλάδας που εγκρίθηκε με στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και την σταθεροποίησή της. Προτείναμε στο Eurogroup, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ένα μεγάλες κλίμακας οικονομικό πακέτο, πακέτο σταθεροποίησης με 110 δισεκατομμύρια ευρώ το Eurogroup, όπου συμμετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών, αποφάσισε βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δύσκολη απόφαση βέβαια, αλλά πολύ σημαντική, ζωτική σημασία απόφαση. Μια υπεύθυνη απόφαση που έπρεπε να ληφθεί. Τώρα τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει πολύ γρήγορα να επικυρώσουν την απόφαση πιστεύω ότι θα μας στηρίξουν στην προσπάθειά μας. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, δεν αγγίζει μόνο την Ελλάδα, έχει να κάνει με τη σταθερότητα ολόκληρης της Ευρωζώνης. Τώρα υπάρχει μια μικρή φωτιά στην Ελλάδα. Πρέπει να φροντίσουμε η πυρκαγιά αυτή να σταματήσει για να μην κάψει και τις υπόλοιπες χώρες. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να είμαστε λαϊκιστές δεν είναι η στιγμή για να προσπαθήσουμε να έχουμε εύκολα κέρδη. Όχι, πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα. Είναι κατά πάσα πιθανότητα το πιο σημαντικό πολιτικό σχέδιο αλληλεγγύης που έχουμε ποτέ, ε, από το οποίο έχουμε ποτέ περάσει. Τώρα για δύο λεπτά λέει ο Πρόεδρος, ο εισηγητής, ο κύριος Ντόιτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και προσωπικώς για τις παρατηρήσεις σας και επιτρέψτε μου να διατυπώσω τρεις ε, συμπερασματικές παρατηρήσεις ύστερα από όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε τόσο καιρό. Είναι γνωστή η φράση ότι για να κάνει κανείς πόλεμο χρειάζεται χρήμα, χρήμα και χρήμα. Για την επίλυση λοιπόν τέτοιων προβλημάτων όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε για τη δημιουργία νέων εργασία, ναι, χρειαζόμαστε χρήματα. Σε πρώτη θέση, σε πρώτη γραμμή χρειάζονται τα χρήματα και είναι πολύ σημαντικό η ΕΤΕΠ να αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά για να βοηθήσει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ή να διαφυλάξουμε τι εργασίε που έχουμε. Μα έχει σταθεί πολύ τιμιαρογός όλα αυτά τα χρόνια η ΕΤΕΠ. Ήταν πολύ σημαντικέ οι επεμβάσει, παρεμβάσεις των συναδέλφων. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το ότι εντοπίστηκε το ότι πλήττονται ιδιαίτερως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την κρίση που διερχόμαστε σήμερα και ιδιαίτερος το ότι έχει και τις εξωτερικές δραστηριότητες της να αναπτύξει η Επίσης κάποιοι συνάδελφοι μίλησαν για την εντολή της και τη σημασία να προσφερθεί ενίσχυση και στα κράτη, τα γειτονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερως δηλαδή την Ουκρανία και τα κράτη της Βαλκανικής. Επιτρέψτε μου επίσης, στο τέλος αυτής της ε, δουλειάς, αυτής της παρεμβάσεως, να απευθυνθώ στους κύριους Κλάιναν και Ντεπίτο, πολύ σημαντικούς εταίρους στις προσπάθειές μου. Με βοήθησαν ιδιαίτερως στην σύνταξη αυτής της έκθεσης. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστώ και τους συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ντόιτς, λέει ο πρόεδρος. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και το έργο σας στην έκθεση αυτή. Το λόγο ξαναζήτησε ο κύριος Χανς Πέτερ Μάρτιν για προσωπικές συνήξεις. Yeah. Πρόεδρε, Προηγουμένως, ο συμπατριώτης ο κύριος Μέλτσερ αναφέρθηκε σε εσά, ε, στο, στο, ιστορικό σας, ε, στη συμπεριφορά σας και με βάση το άρθρο 151 έχετε δικαίωμα απάντησης. Τέτοιου είδους προσωπική υπενιγμή όμως και τέτοιες συζητήσεις δεν μπορούν να μετατραπούν σε μάτς πινκ pong στο ένα θα υπενίστε τον άλλον και ο άλλος θα ανταπαντά και θα έχουμε συνέχεια στιχομηθίε. Να τελειώσει αυτό το θέμα. Ένα λεπτό έχετε κύριε Μάρτι για να απαντήσετε. Αλλά παρακαλώ θερμά να περιοριστείτε σε αυτά που προβλέπει το άρθρο 151 του κανονισμού και στο λεπτό πάνω, λεπτό και ένα δευτερόλεπτο θα πενεργοποιήσω το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Είναι θλιβερό το ότι υποχρεούται η Ολομέλεια να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι ο κύριο Μέλτσερ ε, ψεύστη εδώ μέσα. Ναι, ήταν εκείνο ο οποίο με απεκάλεσε ψυχασθενή. Είναι πολλέ οι περιστάσει πέρσι όπου με παρέπεμψε σε ψυχιατρική κλινική. Είναι αυτή η πολιτική των Ναζί. Άλλωστε το είπε και ο πρόεδρο τη Ελληνική Ομάδα πέρυσι ότι πρόκειται για ομάδα τη οποία ηγείται ο κ. Μιόλτσερο, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην ιδεολογία του νεοναζισμού. Έτσι λοιπόν, χρηματοπιστωτική κρίση, οικονομική κρίση, ο οικονομικό πόλεμο, αν θέλετε, ναι, μα απασχολούν, αλλά πρέπει να δούμε τι συνέπειε έχουν ω προ την παρουσία τη ακροδεξιά στην πολιτική μα ζωή βρίσκονται εδώ είναι ανησυχητικές εξελίξεις και στην Αυστρία και στην Ουγγαρία και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις εξελίξεις. Μάλιστα. Με βάση την ημερήσια διάταξη, από τις 11 θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες.